25 άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε. Απορρίπτεται. Με 9 υπέρ 9 κατά. 26. Τροπολογία 26 άρχεται. Έληξε. Εγκρίνεται με 17 ψήφους και μία αποχή. 27 άρχεται. Έληξε. Απορρίπτεται με 9 υπέρ 9 κατά. Ε, 3 της ΕΚΟΝ άρχεται. Έληξε. Απορρίπτεται με 10, 10 κατά και 8 υπέρ. Της ΕΚΟΝ τροπολογία 4 Άρχεται. Έληξε. Απορρίπτεται με 10 κατά και 8 υπέρ. Τέσσερα, Τροπολογία 4. Άρχεται. Έληξε. Εγκρίνεται με 17 υπέρ και μία αποχή. 5. Άρχεται. Έληξε. εγκρίνεται με 17 υπέρ και μία αποχή. 6 άρχεται, έληξε, εγκρίνεται με 18 ψήφους. Προφορική τροπολογία 3 άρχεται, έληξε, εγκρίνεται με 18 ψήφους. Η 7 καταπίπτει 1. Άρχεται. Έληξε. Εγκρίνεται με 16 υπέρ 2 κατά. 2. Τροπολογία 2 άρχεται. Έληξε. Απορρίπτεται. 9 υπέρ 9 κατά. 3. Άρχεται. Τροπολογία υπερθμών 3. Έλξη. Όχι, κάποιο λάθο έγινε. Λοιπόν, παραλαμβάνω την ψηφοφορία. Τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Έλξε. Εγκρίνεται με 17 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 4. Προφορική. Άρχεται. Έλξε εγκρίνεται με 18 υπέρ. Και θέτουμε σε ψηφοφορία ε, το συνολικό ψήφισμα όπως διαμορφώθηκε μετά την ψηφοφορία. Άρχεται. Έληξε. Εγκρίνεται με 17 ψήφους υπέρ και μία αποχή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναδούμε, θα τα ξαναβούμε στην επόμενη συνεδρία στις 22 Μαρτίου στις 3 το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Ναι, και ωράριο... 12.30. Allora la lettera la prepara lei, mi sembra, poi ci vediamo dopo.